Τα πρακτικά της συνεδρίασής μας θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή μας εάν δεν υπάρχουν καθόλου ε, αντιρρήσεις. Τα ψηφίσματα αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί θα διαβιβαστούν στους αρμόδιους.